Okay, Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε αργήσει ήδη κάποια λεπτά να φροντίσουμε ο χρόνο που καθυστερήσαμε να αφαιρεθεί από το δικό μου χρόνο ομιλία. Ε, χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι εδώ σήμερα και ε, προεδρεύω αυτή τη ε, ακρόαση. Θα ήθελα ιδιαίτερω να καλωσορίσω από πλευρά τη Επιτροπή μα τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίο έχει διοριστεί για Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων. Κάποιοι από εσάς ήσασταν εδώ χθε το βράδυ. Για όσου ε, δεν είσαστε εδώ πέρα, θα ήθελα να εξηγήσω εκ νέου τη διαδικασία. Το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον ε, άρθρο 118 και παράρτημα 16 του κανονισμού, προετοιμάζει τι ε, ακροάσεις αξιολογώντας όλους τους υποψηφίους ε, επιτρόπους βάσει της γενικών τους ικανοτήτων, τη δέσμευσή τους σε ευρωπαϊκά ζητήματα και της προσωπικής τους ανεξαρτησίας. Επίσης, το Κοινοβούλιο αξιολογεί την κατανόηση του χαρτοφυλακίου του υποψηφίου και τις ε, επικοινωνικές του ικανότητες. Και αυτό το σκοπό λοιπόν εξυπηρετεί η σημερινή ακρόαση, να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Να σας ενημερώσω ότι η ακρόαση αυτή μεταδίδεται ε, ζωντανά στο, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Europe by Satellite. Καλώς ορίζουμε λοιπόν και όσους μας παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου ή μέσω του Europe by Satellite, μέσω δορυφόρου. Ε, οι μαγνητοσκοπήσεις επίσης θα διατεθούν μετά την ακρόαση από όσους το ζητήσουν. Για την σημερινή ακρόαση έχουμε διερμηνία σε 23 γλώσσες. Όλοι έχουν χρονική πίεση, αλλά σας παρακαλώ να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα για να μπορούν να σας παρακολουθούν και οι διερμηνείς. Είναι μάλιστα σήμερα και η Διεθνή ημέρα της μετάφρασης. Άρα ευχόμαστε σε όλους του διερμηνείς μας ε, καλή ημέρα της μετάφρασης και χαιρόμαστε πολύ που τους έχουμε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα και από εμάς. Έχουμε αποστείλει κάποιες γραπτές ερωτήσεις στους υποψηφίους, στον υποψηφίο επίτροπο και έχει απαντήσει. Έχετε αντίτυπα των απαντήσεων και διατίθενται άλλωστε και στην αίθουσα για, του, για τους βουλευτές. Να σας εξηγήσω τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Θα ξεκινήσει ο Κριστιλιανίδης με μία δήλωση 15 λεπτών κατά ανώτατο όριο. Και το βασικό τμήμα της ακρόασης θα αποτελείται, όπως και χθες το βράδυ, από 45 ερωτήσεις. Στον πρώτο γύρο κάθε πολιτική ομάδα θα έχει μία ερώτηση ενός λεπτού και ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει 1,5 λεπτό για να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Μετά την απάντηση του υποψηφίου επιτρόπου. Θα υπάρχει ενδεχομένω ε, δεύτερη ερώτηση, υπερέτηση για 30 λεπτών και απάντηση ενό λεπτού. Τέσσερα λεπτά λοιπόν σύνολο για τον πρώτο γύρο. Όλε οι υπόλοιπε ερωτήσει θα διαρκέσουν ε, τρία λεπτά σύνολο. Μία, ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση. Συνάδελφοι, παρακαλώ να έχετε υπόψη τα χρονικά περιθώρια, το χρονικό πλαίσιο, γιατί δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τον προβλεπόμενο χρόνο. Επίσης θα έχουμε ερωτήσεις από τις δύο επιτροπές που έχουν προσκληθεί στην ακρόαση γιατί εμπίπτουν ε, στον τομέα των αρμοδιτήτων τους ε, το χαρτοφυλάκι του υποψηφίου επιτρόπου είναι η Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημοσίας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και μετά θα ανοίξει η συζήτηση για ερωτήσεις από τις πολιτικές ομάδες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα. Κυρία Στυλιανίδη, έχετε το λόγο για 15 λεπτά maximum. Σας ευχαριστώ πολύ.